A ver, pueden sentarse todos y callarse los que están en conversaciones aquí. Μπορείτε σας παρακαλώ να σταματήσετε τα πηγαδάκια εδώ μέσα στην αίθουσα και να καθίσετε. Κυρία Ντότ, σας παρακαλώ. Mrs. Dodds, please, can you take a seat, please? Ε, ε, παρακαλώ, καθίστε. Κύριε Ρόντου, νομίζω ότι μπορείτε να ξεκινήσετε τώρα. Ich glaube, jetzt äh, ist es etwas ruhiger geworden und... Ναι, ναι, έχει μεγαλύτερη ησυχία τώρα και μπορώ να αρχίσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Πρόεδρο για το διάλειμμα αυτών των δύο λεπτών. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ χρήσιμο. Αγαπητοί συνάδελφοι, για πρώτη φορά παρουσιάζω σήμερα τον βασικό κανονισμό. Θα περιοριστώ στο τμήμα 1 στόχους δηλαδή και το MSI. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εκείνους που τις τελευταίες μέρες, τις τελευταίες εβδομάδες ε, μας τηλεφωνούν, θέλουν να συζητήσουν μαζί μας, μας στείλουν ε, ηλεκτρονικά γράμματα και όλους τους συναδέλφους επίσης που έδρασαν για την προετοιμασία αυτού του βασικού κανονισμού ιδιαίτερες ευχαριστήσεις. Νομίζω ότι το τελικό αποτέλεσμα θα είναι ένα πολύ καλό κανονισμό. Ε, θα πρέπει να δούμε του γενικού στόχου. Η κυρία Πατράου Νέβες προετοίμασε το βασικό έγγραφο για το ΒΕΣΤΕ και υπήρχε μεγάλη συζήτηση κατά πόσο θα πρέπει να έχουν ε, την ε, πρωτοκαθεδρία η οικολογική ε, στόχη και όχι η κοινωνική και οικονομική. Νομίζω θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί γιατί αλλιώς έχουμε μία ψευδοσυζήτηση γιατί νομίζω ότι η κοινωνική και η οικονομική στόχοι μπορούν να επιτευχθούν μόνο εάν είναι οικολογικά βιώσιμα τα αποθέματα. Είναι σαφές και τονίζεται προστάχης ότι η πολιτική ας πούμε, είναι υπέρ των ανθρώπων και θέλουμε οπωσδήποτε μία ηλιή αγία. Αλία, συγγνώμη. Όλα λοιπόν είναι ισότιμα στη συζήτηση. Θέλουμε υγιείς θάλασσες και θέλουμε και υγιή ε, αποθέματα ε, λιθμάτων. Όλα αυτά είναι προς όφελος των ανθρώπων, αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός. Η πρόταση της ε, Κομισιόν ε, μ' αρέσει όσον αφορά την ε, πολιετή της κατεύθυνση και μακροπρόθεσμα συμπίπτουν όλοι οι στόχοι. Σχεδόν. Σχεδόν γιατί η αξιολόγηση των επιπτώσεων δείχνει ότι υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά την οικονομική αποδοτικότητα και την κοινωνική πτυχή. Η παραδοσιακή αλληλεία επιτρέπει υψηλά επίπεδα απασχόλησης, αλλά δεν είναι οικονομικά αποδοτική. Και ε, επίσης, ε, ε, αν δεν έχουμε υγιή α, το ε, υγιή παράκτια, ε, απειλείται και ο τουρισμός. Μετά. Όλοι συμφωνούν ότι θα ήταν καλό τα αποθέματα, τα λεφτικά να είναι κατά δυνατόν υψηλά. Αυτό όμως είναι ε, γελίο, γιατί καταφέραμε στην κατάσταση που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή να μειώσουμε τα αποθέματα. Και νομίζω αυτό δεν είναι προς όφελος ουδενός. Και είμαι πεπισμένη ότι οι στόχοι του MS2 θα πρέπει να είναι αυστηροί και με μεγάλη ακρίβεια διατυπωμένοι. Αλλιώς δεν θα πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Οποιαδήποτε διατύπωση ασαφής θα τύχει εκμετάλλευσης. Θα πρέπει να δούμε ποιος είναι ο ορισμός του MSY. Υπάρχει ορισμός της ΦΑΟ που αποκρίνει από αυτό που αναφέρεται στο άρθρο 5. Επίσης θα πρέπει να λύσουμε προβλήματα πράκτικες. Το πρώτο είναι πώς θα επιτευχθεί ο στόχος του 2015. Το δεύτερο, κατά τη γνώμη μου, είναι το πρόβλημα στη μεικτή αλία. Και το τρίτο πρόβλημα είναι στην ε, ε, ακτή. Δηλαδή, αρχίζω με το πρώτο σημείο, 2015. Για ορισμένα από το ξέρουμε όλοι, που χρειάζονται μεγάλα χρονικά διαστήματα για να ανανεωθούν, είναι ε, βιολογικά αδύνατο να πετύχουν αυτούς τους στόχους. Όμως, και το λέω αυτό ξεκάθαρα, αυτό δεν είναι λόγος να αποκλίνουμε από τον στόχο μας. Ε, θα πρέπει ίσως για τα αποθέματα αυτά να έχουμε ενδιάμεσους ε, στόχους. Εάν αυτό το MSY, το όριο μέγιστη διαρκούς απόδοση δηλαδή, δεν επιτυγχάνεται, θα πρέπει ίσως να μειωθεί. Καταρχήν, στο βασικό κανονισμό θα πρέπει να είναι απόλυτα σαφές ποια είναι η διάσταση του MSY που εννοούμε βιομάζα, ελαφρά βιομάζα ή θνησιμότητα αλληλευτική. Gemischten Fischereien. Einige, mit denen ich ε, ορισμένοι με οποίους συζήτησα, το έξω και εδώ, ε, λένε ότι αν υπάρχει μεικτή αλία, τότε είναι αδύνατο να υπάρχει MSY. Εγώ λέω ότι αυτό δεν είναι σωστό, γιατί τα αποθέματα του MSY μπορούν να επιτευχθούν. Βέβαια υπάρχουν ε, διακυμάνσεις. Αλλά αυτές κινούνται ε, σε ένα μέσον όρο. Εγώ θα έλεγα και έχω να σας το προτείνω ότι το πιο αδύναμο μέλος στην αλυσίδα τη διατροφική στη θάλασσα είναι εκείνο που ορίζει. Γι' αυτό θα πρέπει να βρεθεί μία δυνατότητα να αυξηθεί η επιλεκτικότητα της αλίας. Μόνο έτσι ωφελούνται και οι αλίες από τα μεγαλύτερα αποθέματα. Και νομίζω ότι αυτό είναι ο στόχος μας. Συμφωνούμε σε αυτό. Ένα από τα σημεία που πρέπει να βελτιώσουμε είναι κατά πόσον αυτός ο στόχος του MSY είναι δεσμευτικός για τις ετήσιες ποσοστώσεις των κρατών μελών. Η Κομισιόν θέλει να έχει πολυετή στόχους. Ξέρουμε όμως από τις ε, συζητήσεις του παρελθόντος ότι τα πολυετή σχέδια δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να υιοθετηθούν. Και γι' αυτό θα πρέπει το Συμβούλιο και χωρίς πολυετής ε, ε, προτάσεις να μπορεί να εφαρμόσει αυτό ε, το κανισμό, κανονισμό, ώστε να επιτευχθούν οι δικοί μας στόχοι. Μετά, τι θα κάνουμε το μεσβαί αν δεν έχουμε επαρκής, επαρκή στοιχεία. Ο βασικός κανονισμός θα πρέπει να υποχρεώνει σε περισσότερα πράγματα τα κράτη-μέλη, ώστε να ε, μεταβιβάζουν τα στοιχεία τους. Καμιά φορά δεν ε, υποβάλλονται ούτε οι στατιστικές, μου είπαμε. Αυτό είναι σκανδαλώδες. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε κυρώσεις και ε, οθήσεις που θα οδηγήσουν στο σωστό στόχο. Επίσης, το άρθρο 4 είναι σημαντικό να υπάρχουν οι αρχές για την καλή λήψη αποφάσεων. Είναι σαφές ότι αυτά τα σημεία θα πρέπει να περάσουν στο πνεύμα εκείνο που θα λάβουν την απόφαση, ιδίως το α όσον αφορά την οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων των διαφόρων επιπέδων, β η επιστήμη σαν βάση και γ οι μακροπρόθεσμες προοπτικές και δ πλήρη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων ομάδων. Αυτά μου φαίνονται πάρα πολύ σημαντικά. Και θα πρέπει εδώ να εκμεταλλευτούμε τα μέσα που υπάρχουν, όπως την Επιτροπή Τεχνολογίας και Επιστήμης και ε, αυτά μπορούν να μας στηρίξουν. Για μένα είναι σημαντική αρχή ότι πάντα θα πρέπει να σκεφτούμε να μειώσουμε τη γραφειοκρατία και να αποφύγουμε την περιττή γραφειοκρατία. Ξέρω ότι αυτό είναι κάτι που συζητιέται παντού. Ε, αυτό είναι κάτι που το ζητάμε εδώ και πολλά χρόνια, δεν το πετυχαίνουμε, αλλά τώρα έχουμε πάλι μια ευκαιρία να το κάνουμε. Και θα πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε να έχουμε, εν τελευταία αναλύση, λιγότερη γραφειοκρατία. Γιατί αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι απαράδεκτο για πολλούς. Όσον αφορά προσωρινούς ε, κανόνες, ε, μπορούμε να το έχουμε, αλλά κατά τα άλλα είναι καλύτερο να έχουμε ε, οθήσεις και όχι χιλιάδες σελίδων κανονισμού. Αν δεν αρκούν τα κίνητρα, χρειαζόμαστε βέβαια κάποιες άγουσες. Εγώ δεν θέλω αναρχία στη θάλασσα, ούτε και εσείς φαντάζομαι θα το θέλετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Merci, Madame Ευχαριστώ, ε, Πρόεδρε. Επιτέλους, περάσαμε στο ψαχνό. Ευχαριστούμε την κυρία Ροντούστ. Βέβαια καλή τύχη κυρία Ροντούστ, διότι το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, δεν ε, ικανοποιεί τους πάντες, τουλάχιστον όχι όλα τα σημεία του όπως βλέπουμε. Ε, έχουμε μέσα σε αυτόν τον κανονισμό του μελλοντικού στόχου τη κοινή ελευθερική πολιτική. Είναι οριζόντιο το θέμα σχετικά με τι διάφορε πολιτικέ ε, τώρα τη ε, Ένωση και συγκεκριμένα η περιβαλλοντική πολιτική. Νομίζω ότι είναι ικανοποιητικά τα στοιχεία. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εντάξει είναι σημαντικό ο γενικό στόχο τη κοινή αλληλευτική πολιτική, αλλά εξίσου σημαντικό είναι και ο κοινωνικό πυλώνα. Ε, ο περιφερειακός πυλώνα. χρειαζόμαστε μια ρεαλιστική πολιτική ούτω ώστε να λάβουμε ε, υπόψη ε, όλους τους τομείς ε, της αλίας. Ε, θα πρέπει να βελτιώσουμε τις συνθήκες εργασίας ε, των Αλίων, το εισόδημά τους, το, την κατάσταση την οποία ζουν. Σχετικά με τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση και το στόχο για το 2015, νομίζω, θα πρέπει να ε, τηρήσουμε τις δεσμεύσεις που αναλάβαμε στο Johannesburg και στην Κογιάννα. Για το 2015 πάντως εμένα δεν μου φαίνονται ρεαλιστικοί οι στόχοι. Θα πρέπει αναλύευμα να αποφασίσουμε, αναπόθεμα να αποφασίσουμε τη μέγιστη απόδοση ε, μέσα σε ένα πολιετέ ε, πλαίσιο, λαμβάνοντας υπόψη και το μακροπρόθεσμο αντίκτυπο αυτών των μέτρων. Ε, Ούτω ώστε να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι τη κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Για τις απορρίψεις που είναι το Δεύτερο αμφιλεγόμενο σημείο στη συζήτηση, η σταδιακή μείωση των απορρίψεων είναι κάτι το ευκταίο και κάτι το απαραίτητο. Αλλά η γενικευμένη μείωση των απορρίψεων, όπω προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν συνιστά ρεαλιστική πρόταση, κατά τη γνώμη μου. Υπάρχουν πολλέ αιτίε για την απόρριψη μη προσαρμοσμένα τεχνικά μέτρα, ε, και ηχθιδίων κτλ. Αναπόθεμα και πάλι πρέπει να προσαρμόσουμε τα μέτρα. Ε, μπορούμε να γενικεύουμε τα μέτρα, να μειώσουμε γενικότερα τι απορρίσει. Ε, ε, είναι σημαντικό να έχουμε προληπτικά μέτρα, όχι μόνο να επιδιορθώνουμε τι ζημιέ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόνο μέτρα ε, επανόρθωσης κατάσταση μας προτείνει και όχι προληπτικά. Σχετικά με τις μεταβιβάσιμες ποσοστώσεις, εδώ ε, σας ξαφνιάσω να σας πω ότι είμαι κάθετα αντίθετος, γνωρίζετε τη θέση μου. Δεν είμαι υπέρ της υποχρεωτικής ε, θέσπισης ενός μεμονωμένου ε, συστήματος ανταλλαγής ε, ποσοστώσεων που με συγκεκριμένο αντίτυπο, διότι έτσι θα ευνοηθεί η κερδοσκοπία και η υπερβολική συγκέντρωση των ε, ποσοστώσεων ε, δημιουργώντας μια αγορά δικαιωμάτων, αλληλευτικών δικαιωμάτων. Εάν ε, έχουμε αυτό το σύστημα για τη βιομηχανική λία, ήταν μια υπόθεση, σίγουρα αργά ή γρήγορα θα, εφαρμοστεί και για την εραστεχνική αλία όπως έγινε στην Ισλανδία. Πρέπει να απαγορεύσουμε θέσπιση αυτού του συστήματο των μεταβάσιμων ποσοστώσεων για τη διακυβέρνηση και το άρθρο 4 προτείνεται ενεργό συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων μερών από τη σύλληψη μέχρι την έγκριση και την εφαρμογή των μέτρων. Ε, καλή ιδέα, αλλά αυτό δεν φαίνεται με σαφήνεια στον κανονισμό. Θα ήθελα να ενισχυθεί πάρα αυτά το περιφερειακό επίπεδο, η περιφερειοποίηση στο κείμενο δεν φαίνεται, ενώ ήταν στην πράσινη βίβλο, όπως την παρουσίασε η Επίτροπος εδώ στο Κοινοβούλιο, όμως δεν το βλέπουμε σε αυτό το έγγραφο. Πρέπει να ενισχύσουμε την περιφερειακή διάσταση, αλλά στην εφαρμογή επίσης για να λάβουμε υπόψη τις ιδιαιτερότητες των διαφόρων ε, λεκανών αλίας ε, μέσω, αυτών των περιφερειακών ε, γνωμοδοτικών συμβουλίων που θα πρέπει να εργαστούν, να συνεργαστούν μάλλον στενά με τα κράτη-μέλη. Πιστεύω ότι θα γίνουν έντονες συζητήσεις. Δεν νομίζω ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία, ούτε νομίζω ότι η μεταρρύθμιση θα ικανοποιεί ε, όλα τα μέλη τη Επιτροπής. Θα ήθελα να διευκρινίσω το εξή. Έχουμε αποφασίσει ότι σε κάθε συνεδρίαση θα μιλάμε για συγκεκριμένα θέματα και όχι να μιλάμε γενικώ ε, για όλη τη μεταρρύθμιση τη κοινή αλληλευτική πολιτική. Σα παρακαλώ λοιπόν να τηρήσετε αυστηρά αυτό τον κανόνα και να περιοριστείτε μόνο στα θέματα που θα συζητήσουμε σήμερα και μην αρχίσουμε τι γενικόλεγε συζητήσει γιατί αλλιώ δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε συγκεκριμένα για κάθε θέμα σε κάθε συνεδρίαση. Σα παρακαλώ να περιοριστείτε στα άρθρα 1 έω 5 του κανονισμού, τίποτα άλλο. Δεν συζητάμε ούτε περιφερειακέ οργανώσει ούτε τίποτα άλλο σήμερα. Κύριε Στίβενσον, ελπίζω εσεί να τηρήσετε αυτά που είπαμε και έχουμε καθορίσει για σήμερα. Παρακαλώ. Sorry, chairman, after Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Μετά από την επίπληξή σας δεν ήμουν βέβαια αν έπρεπε να μιλήσω. Δεν πειράζει, μπορούμε να προχωρήσουμε και χωρίς εσά λέει η Πρόεδρος. Το μόνο που ήθελα να πω είναι το χρονικό όριο της όλης κατάστασης. Το ανέφερε και η κυρία Ρόντες, το ανέφερε και ο κύριος Καντέκ ε, το MSY, τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Κοιτάμε την εφαρμογή ε, του όλου πακέτου μεταρρύθμισης και θέλουμε να ξεκινήσει 1η Ιανουαρίου του 2013. Αποκλείεται να τα καταφέρουμε. Η πιο γρήγορη πρώτη ανάγνωση μέχρι τώρα από τότε που τέθηκε σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας ήταν 18 μήνες. Εάν δημοσιευθούν λοιπόν ε, τα πράγματα όπως δημοσιεύθηκαν στις 13 Ιουλίου ε, είμαστε σαφώς μετά από το 2013 χωρίς να καν να διανοηθούμε συμφωνία σε δεύτερη ανάγνωση. Θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι να μην ε, περάσουμε και στο 2014 γιατί την 1η Ιανουαρίου του 2014 δεν θα έχουμε πλέον νομική βάση και επομένω καταστρεπτική η κατάσταση. Θα πρέπει να είμαστε λοιπόν πολύ προσεκτικοί ε, οτιδήποτε έχουμε να συζητήσουμε οποιασδήποτε νομικής φύσης διαφορές μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων δεν θα πρέπει να ε, οδηγηθούν και να παρατεθούν πέρα από το 2013. Όλα αυτά βέβαια έχουν επιπτώσεις για το MSY όπως σα έλεγα. Το αρχικό χρονοδιάγραμμα ε, ήταν γελίο. Ξέρω ότι είχαμε τη συμφωνία του Johannesburg, αλλά ακόμα και αν κλείσουν όλες οι δυνατότητες αλληλείας ε, στην Ευρώπη, αποκλείεται να πετύχουμε το MSY που θέλουμε μέχρι το 2013. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Ε, υπάρχουν συνέπειες και για το χρονοδιάγραμμα για τις απορρίψεις, αναείδος. Δεν μπορούμε να επιτύχουμε ούτε αυτά τα χρονοδιαγράμματα και δεν ε, ε, πίστεψα ποτέ βέβαια εγώ ότι υπήρχε δυνατότητα να καταφέρουμε τους στόχους που είχαμε θέσει, αλλά θα ήθελα να ακούσω και την άποψη της κυρίας Ρόνταστε. Τι νομίζετε ότι πρέπει να κάνουμε με το χρονοδιάγραμμα, γιατί αυτό θα έχει επιπτώσεις και στη δική μου την έκθεση για την ε, κοινή οργάνωση αγοράς. Ευχαριστώ κύριος Ντέιβις. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα για τον ορισμό του MSY εντάξει, καλή η ερώτηση, γιατί υποθέτω ότι υπάρχουν πολλοί ορισμοί. Προφανώ έχει έναν κατά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ίσω ε, προ το τέλο συζήτηση να διευκρινίσει τι προθέσει τη. Αλλά μην ξεχνάμε ότι υπάρχει η Διεθνή Συμφωνία του Γιωχάνεσμπουργκ, οπότε πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι συμμορφωνόμαστε με τα πρότυπα που έχουν εγκριθεί σε άλλα φόρα. Δεύτερον, Ε, σχετικά με τη δυνατότητα επίτευξη του στόχου. Εγώ ήμουν στην, ε, ε, στο, στο Johannesburg και η κυρία Βίξτρομ ήταν εκεί και έκανε την εξαγγελία στο, στη συνέντευξη τύπου. Τέλος πάντων, στο μεταξύ εγκρίθηκε και η συνθήκη της Λισαβόνας είναι ελεύθερο να κινηθεί το κοινοβούλιο, πάντως τα κράτη-μέλη δεν τα έχουν καταφέρει καλά σε σχέση με την τήρηση των διεθνών δεσμεύσεών τους. Στην ουσία δεν γίνεται να επανέλθουν τα αποθέματα στο επιθυμητό επίπεδο στο χρόνο που μας μένει. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να έχουμε μεγάλες φιλοδοξίες, να ασκήσουμε πίεση, ε, να θέτουμε σκληρούς φιλόδοξους στόχους, ε, ε, ακόμη και αν σημειώνονται παρεκτροπές Ε, ε, δεν μπορούμε δηλαδή να ρίχνουμε μια ιδέα και να λέμε «Α, δεν τα καταφέρουμε μέχρι το 2015, ας μετατοπίσουμε τη ημερομηνία το 2023». Αυτό το ε, MSY μπορεί να θεωρηθεί όχι μόνο ως μέγιστη αλλά ως και ελάχιστη απόδοση. Δεν ε, αρκεί αυτό. Ε, Εμεί δεν θέλουμε μόνο να καταπολεμήσουμε την υπερα, υπεραλίευση. Θέλουμε, εγώ θέλω να έχουμε τα αποθέματα όπως παλιά. Θέλω να μειώσουμε τις αγωγές ψαριών, να αποκαταστήσουμε τα εισοδήματα των ψαράδων πρέπει να κάνουμε την υπέρβαση πέραν της ε, ανώτατης ε, μέγιστης, της μέγιστης συγγνώμη, ε, βιώσιμης απόδοσης. Ε, κυρία Λέβιν, ευχαριστώ, ευχαριστώ την κυρία Ρόντους ε, για την εισαγωγή της. Ε. Έχω διάφορες παρατηρήσεις. Λοιπόν, για το MSY, φυσικά όπως είπε και ο κύριος ε, Στίβενσεν, δεν θα μπορέσουμε να επαναφέρουμε τα αποθέματα ως προς τη βιομάζα ε, μέχρι το 2015. Υπάρχουν δύο τρόποι μέτρησης για το MSY. Η πρώτη είναι για τη βιομάζα και η άλλη ε, σχετίζεται με θνησιμότητα των ψαριών. Υπάρχει και το F ε, το FMSY, το δεύτερο, μπορούμε να το εφαρμόσουμε αύριο. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε μέχρι το 2020 ή οποιαδήποτε άλλη χρονιά, αλλά ε, μιλάμε για ένα ποσοστό υπερεκμετάλλευση, ε, το οποίο είναι άμεσα εφαρμόσιμο. Θέλω να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όταν μιλάτε για την μέγιστη βιώσιμη απόδοση, δεν πρέπει να διευκρινίσουμε τι ακριβώς εννοούμε. BMSY ή FMSY, για ποια από τις δύο κατηγορίες. Ε, γιατί, γιατί η δεύτερη σε σχέση με τη θνησιμότητα είναι άμεσα εφαρμόσιμο το ποσοστό και αυτό πρέπει να κάνουμε εξάλλου. Άλλη παρατήρηση. Αυτή η λέξη above, υπέρ, χρησιμοποιείται μέσα στο κείμενο υπέρ της ε, μεγίστης απόδοσης ε, για ε, ότι πρέπει οι πληθυσμοί αυτών των ειδών να παραμένουν ε, άνω υπέρ αυτού του, αυτού του επίπεδου του MSY. Όμως τα είδη δεν ζουν απομονωμένα. Ξέρετε, ε, υπάρχει ε, στενή επαφή, υπάρχουν οι θηρευτές, υπάρχουν ε, τα, τα θυράματα και χρειαζόμαστε ε, κάποιες εγγύησεις ε, για τα αποθέματα, γιατί δεν γίνεται να ε, ε, εκμεταλλευόμαστε κάθε είδος απομονωμένα και να παίρνουμε τη μέγιστη απόδοση ανά είδος. Είναι αδύνατον αυτό, οπότε θα πρέπει να ορίσουμε ανώτερα επίπεδα. Αφήστε που πρέπει να λάβουμε υπόψη το ρόλο που παίζουν τα διάφορα είδη για, την, για να παραμένουν υγιεί τα οικοσυστήματα. Ε, είναι μια άλλη λογική. Δεν υπάρχει μόνο η λογική της ε, ε, υπερεκμετάλλησης, υπάρχει και η λογική των οικοσυστημάτων. Αν θέλουμε τα είδη να επιτελούν αυτό το ρόλο τους για να είναι υγιείς οι θάλασσες μας και θα δούμε τα φύκια και τις... Ε, τις μέδουσες να κατακλείζουν τις θάλασσές μας. Πρέπει να αλλάξουμε. Δεν μπορούμε να ακολουθούμε μόνο τη λογική της υπερεκμετάλλευσης. Οπότε Θέλω να είμαστε προσεκτικοί με αυτή τη λέξη above, ε, να παραμένουν τα αποθέματα άνω αυτού του MSY. Προσοχή, στο άρθρο 3 για την απαγόρευση περί απορρίψεων ε, μιλάμε ε, μιλάμε για κατάργηση των ε, μη επιθυμητών ειδών, αλλά για εμπορικά είδη. Ε, παρά είναι περιοριστικό αυτό. Υποθέτω ότι αυτά τα εμπορικά αποθέματα θα καταγραφούν σε ένα κατάλογο. Σίγουρα το σκέφτεται αυτό η Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή. Δε σίγουρα δεν πρόκειται για όλα τα είδη όπου υπάρχουν ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. δεν θα ήταν αντιπαραγωγικό να μιλήσουμε μόνο για ορισμένα είδη και να ε, ε, ξεχάσουμε τα υπόλοιπα. Δεν θα δημιουργηθεί πρόβλημα ελέγχου. Ποια είδη απορρίπτουν, επιτρέπεται να απορρίψουν αυτά τα είδη κτλ. Ε, εγώ πιστεύω ότι χρειαζόμαστε ένα κατάλογο εξαιρέσεων, όπως η Μέδουσες είχε οι χελώνες ε, ή οι καρχαρίες μπορούν να επιζήσουν, ε, να επιβιώσουν μετά από αυτή την εμπειρία της απόρριψης, ε, θα ήταν μια καλύτερη ιδέα μια λίστα εξαιρέσεων ε, δίπλα στην απαγόρευση. Τώρα, ε, για τους στόχους ε, της αλλιευτικής πολιτικής πιστεύω πως είναι εξαιρετικά σημαντικά, σημαντικό αυτό το θέμα και επιτέλους έχουμε την δυνατότητα να διορθώσουμε τα πράγματα, κακώς κείμενα που κοίτα κακώς εδώ και πάρα πάρα πολύ καιρό. με την αξιολόγηση της κοινή αλλιευτικής πολιτικής που έγινε το 1991 ε, όταν το η πρώτη μεταρρύθμιση η πράσινη βίβλος Ευρωπαϊκής Επιτροπής λοιπόν του 1991 ήδη τότε μιλούσε για τους, ε, την ε, ανάγκη να τον στόχο στόχων της κοινής αλληλευτικής πολιτικής γιατί εξαρτάται ήδη από τη διατήρηση των πόρων και πρόκειται για ε, εκ των όνων κάνευ προϋπόθεση. Ε, αυτή ήταν η ανάλυση που είχε κάνει ήδη τότε πριν από 20 χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η πράσινη βίβλος τώρα του 2001 επίσης μιλάει για την έλλειψη ιεράρχης των προτεραιοτήτων σε σχέση με τους στόχους ε, της κοινή αλλιευτικής πολιτικής. Είχαμε και την έκθεση του 2007 το Κοινοβουλίο όπου αναγνωρίζεται ως βασικό πρόβλημα της πολιτικής ακριβώς αυτή η έλλειψη ιεράρχης των προτεραιοτήτων. Το 2008 στην ενδιάμεση αναθεώρηση το ίδιο. Στην Πράσινη Βίβλο του 2009 ε, μιλάμε για σαφείς στόχους ε, των πολιτικών ε, που είναι ένα από τα πέντε διαρθρωτικά προβλήματα της κοινής αλευτικής πολιτικής μάλιστα. Το πρόβλημα είναι ότι αν κάθε φορά κάνουμε πολιτικός προς την επιλογή μας και διαλέγουμε ανάμεσα σε μια μελλοντική ε, ιονή ε, ε, περιβαλλοντική καταστροφή και μια σίγουρη οικονομικοκοινωνική καταστροφή αύριο τι επιλέγετε. Φυσικά θα στραφείτε, θα τζογάρετε και θα στοιχηματίσετε στην μελλοντική ενδεχομένως περιβαλλοντική καταστροφή και να αποφύγετε την αυριανή κοινωνική καταστροφή. Ε, όσοι λαμβάνουν τις οι ε, αποφάσεις εμείς, ε, το Συμβούλιο, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν τις ευθύνες όταν βρίσκονται ενώπιον αυτών των διλημάτων. Υπάρχει ο περιβαλλοντικός στόχος που θα θεωρείται ως προϋπόθεση της οικονομικοκοινωνικής βιωσιμότητας, γιατί πιστεύω ότι όλοι αναγνωρίζουν ότι αυτό ευσταθεί και έτσι θα διαχειριστούμε καλύτερα τα αποθέματά μας για το μέλλον. 68% να σας θυμίσω όλων των αποφάσεων TAC του, του Συμβουλίου ε, αγνοούν τις επιστημονικές συμβουλές τα τελευταία 10-15 χρόνια και κατά μέσο όρο 33, ε, έχουμε 33% υπέρβαση των επιστημονικών συστάσεων ε, σχετικά με τις, τα ανώτατα ποσοστά. Είπα η Αυστραλία και άλλοι μέσα στην ομοθέσια τους για τη διαχείριση των ελληνευτικών μπορούν να αναφέρουν ότι προέχει η περιβαλλοντική ε, βιωσιμότητα. Θέλω να το τονίσω αυτό. Δεν υπήρξε κάποιο πράσινο κίνημα. Ε, είχαμε το νόμο Μάγνουσον Στίβενσον που προέκυψε από τον πρώην πρόεδρο Μπούς δεν ασκήθηκε πίεση από πράσινους Ε, Πάντω ε, ε, παραβιάζει ε, κανεί τον νόμο όταν υπάρχει υπέρβαση σε σχέση με τις επιστημονικέ συμβούλε στην Αυστραλία. Έχουν την ανώτατη οικονομική απόδοση που είναι μια ακόμη πιο προληπτική ε, αρχή σε σχέση με τη δυνατότητα αλίευσης ε, στα ύδατα της Αυστραλίας. Λοιπόν, και η ΕΠΑ και η Αυστραλία φροντίζουν πολύ καλύτερα τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες ε, σε σχέση με το παρελθόν προτού ψηφιστεί αυτή η νομοθεσία. Παρακαλώ να το λάβετε όλοι υπόψη. Είμαστε εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να αντλήσουμε, να μάθουμε από τις εμπειρίες των άλλων να σα πω ότι η κυρία Ρότζος πρέπει να φύγει στις 5 και δεν έχουμε και όλο το απόγευμα στη διάθεσή μα για το θέμα αυτό, δυστυχώ. Η κυρία Ντότζ. Thank you, uh, President. Um, and thank you to Mrs. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ την κυρία ρόντου για τα εισαγωγικά τη σχόλια. Πολύ λίγο θέλω να ε, κάνω κάποια σχόλια. Το θέμα της ε, επιλογή των περιβαλλοντικών στόχων ε, πριν από τα οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα των αλλιών δεν θα πρέπει να υπάρχει. Θα πρέπει να έχουμε την δυνατότητα να λάβουμε υπόψη μας και τα μεν και τα δε και να εργαστούμε και στα δύο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό νομίζω. Δεν θα πρέπει δηλαδή να φέρουμε τα μεν σε ανυπαράθεση με τα δε. Θα πρέπει και τα δύο να θεωρηθούν πάρα πολύ σημαντικά το χρονοδιάγραφα για την επίτευξη του MSY και η ανησυχία ότι δεν θα καταφέρουμε να το πετύχουμε πριν από το 2015, ιδίως για τα μη εγκεκριμένα αποθέματα. Πάνω σε αυτό έχω να πω στη Βόρειο Ιρλανδία προετοιμάζουμε ένα καινούριο σύστημα, ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον σχέδιο για τη συστηματική προσέγγιση διαχείρισης της ε, Ιρλανδικής θάλασσας. Θα χρειαστούμε, θα έλεγα, δύο-τρία χρόνια μέχρι να μπορέσει η προσέγγιση αυτή να προχωρήσει σωστά. Οποιοδήποτε προσέγγιση δηλαδή για το MSY θα πρέπει να είναι σφαιρική και θα ήθελα να ενθαρρύνω τους πάντους να εξετάσουμε την προσέγγιση αυτή σφαιρικά και όχι μεμονωμένα γιατί δεν θα φτάσουμε στο στόχο μας. Είναι και αυτό σημαντικό. Συζητήσατε στη μείωση γραφειοκρατίας και ίσως μου θυμάσαι η Πρόεδρος, εάν πω ότι από τότε που ήρθα στο Κοινοβούλιο, σε οποιαδήποτε επιτροπή και αν ήμουνα, συζητιέται το θέμα της μείωση γραφειοκρατίας. Πολύ καλό αυτό, αλλά δεν το καταφέρνουμε. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να μειώσουμε σε μείωση γραφειοκρατίας χωρίς να μιλήσουμε για πραγματική περιφερειοποίηση της πολιτικής. Θα ήθελα να προτείνω ότι υπάρχουν ορισμένοι στην Κομισιόν, πες να σημειώσει η Κομισιόν, που εξετάζουν το θέμα αυτό και ακούστηκε ότι υπάρχουν κάποιες εντάσεις στην Κομισιόν όσον αφορά την υπερπεριφερειοποίηση του θέματος. Αλλά δεν θα μπορέσουμε ποτέ να μειώσουμε γραφειοκρατία αν δεν επιτρέψουμε στους ντόπιου να εφαρμόσουν τις τοπικές αποφάσεις. Και επίσης, η μείωση της γραφειοκρατίας σημαίνει ότι λαμβάνονται υπόψη ανησυχίε των Ελλήνων. Εμείς στην Επιτροπή μας ούτε καν συζητάμε τα νέα τεχνικά μέσα συντήρησης που πρόκειται να εφαρμοστούν από ό,τι κατάλαβα μετά τα Χριστούγεννα όσον αφορά την επιλογή των εργαλείων ε, λίας Και οπωσδήποτε οι αλίες ξέρουν πολλά πράγματα και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις απόψεις τους για να δούμε πώς θα έχει επιπτώσεις αυτό στην αλία. Ευχαριστώ. Εγώ τα λέω για να έχουμε μια σειρά, αλλά τέλος πάντων ε, συζητήσουμε ό,τι θέλετε. Εδώ έχουμε καθορίσει κάποιους όρους και πρέπει να τους ακολουθήσουμε. Ο κύριος Χάκτον. Um, um, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να τηρήσω αυτά που υποτίθεται ότι συζητάμε. Όπως και ο κύριος Καντέκ, ε, θεωρώ ότι θα πρέπει να ακούμε τις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης και χαίρομαι που ο κύριος Καντέκ ζήτησε να ενισχύσουμε την αρχική διάσταση. Μας ενδιαφέρουν τα θέματα της περιφερειακής διάστασης. Στο άρθρο 4 αναφερόμαστε στην κοινή αλληλευτική πολιτική που διέπεται από τις ακόλουθες αρχές χρηστής διακυβέρνησης και έχουμε το σαφή ορισμό των ευθυνών σε ονοσιακό εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο πρώτο-πρώτο. Κατά την άποψή μου δεν έχουμε αρκετή σαφήνεια σε αυτό το τομέα της διακυβέρνησης και δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να ξεκινούμε αυτή τη μεγάλη αναθεώρηση ενός τομέα πολιτικής στον οποίο όπως όλοι αναγνωρίζουμε έχουμε αποτύχει και δεν έχουμε σωστή διαχείριση των ελευτικών αποθεμάτων στα ευρωπαϊκά ύδατα, διότι νομίζω ότι τα θέματα της χρηστής διακυβέρνησης είναι μεταξύ των βασικών αρχών που μας οδήγησαν στην αποτυχία αυτών των στόχων. Και στο άρθρο 4 Αναφέρεται και η ευρεία συμμετοχή των ενδιαφερομένων σε όλα τα στάδια. Αναφέρεται η πρωταρχική ευθύνη του κράτου σημαία. Αναφέρεται η συνοχή με την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική, ε, η οποία σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βοηθά τα κράτη-μέλη και τις ε, ε, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα για να μπορούν να λειτουργούν σωστά. αν θέλουμε να συνεχίσουμε μια κοινή ελευτική πολιτική με ίση πρόσβαση στα ύδατα και στους πόρους και εάν, όπως λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα ε, και γι' αυτό ακριβώς μας λέει ότι δεν μπορεί να προτείνει τόση αποκέντρωση όσο θα θέλαμε. Δεν λέει όμως ότι η αποκλειστική αρμοδιότητα είναι καλή ιδέα και θα μας οδηγήσει σε καλύτερη πολιτική διαχείριση της αλίας, διότι Επειδή όλα αυτά είναι στη συνθήκη, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για να κάνουμε αποκέντρωση τη διαχείριση και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γι' αυτό. Δεν το δέχομαι εγώ αυτό και δεν μπορώ να ακούσω ποτέ κανέναν και από τι συζητήσει ε, που ε, έχουμε εμεί εδώ δεν μπορεί να μας πει πού είναι το καλό στο να έχουμε αποκλειστική αρμοδιότητα ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα θέματα αυτά. Αντιστοίχως δεν άκουσα και κανένα να μας λέει πού είναι το θετικό στο να συνεχίσουμε να έχουμε την, ε, πρόσβαση, την αρχή της ίσης πρόσβασης στους υδάτινους πόρους και στην κοινή αλληλευτική πολιτική. Και να σας πω γιατί. Διότι πιστεύω ότι μεταξύ τους ουσιαστικά υπονομεύουν τις δυνατότητες της ευρωπαϊκής αλληλευτικής πολιτικής για να προσδώσει κίνητρα και τα κίνητρα είναι πολύ σημαντικά όπως λέγει η συγγήτρια, όπως είναι σημαντικοί και οι κανόνες, αλλά αυτές οι ουσιαστικές απειλές και αυτό είναι η συμπρόσβαση σε ύδατα και σε πόρους. Currently have fishing entitlements in, say, the North Sea δεν έχουμε τόση αποκέντρωση όσο θα έπρεπε να έχουμε και έχουμε και κοινά αλληλευτικά δικαιώματα τα οποία θα έπρεπε να έχουν αποτελέσματα. Κάποια στιγμή στο μέλλον η κοινή αλληλευτική πολιτική θα λέει ότι θα πρέπει να υπάρχει ίση πρόσβαση σε ύδατα και πόρους. Πού είναι λοιπόν τα κίνητρα για το μακροπρόθεσμο όφελος πώς μπορούμε να έχουμε μακροπρόθεσμο όφελος ε, για τη διατήρηση των αποθεμάτων και ποιοι είναι αυτοί που έχουν να κερδίσουν για τη διατήρηση ε, των ε, δικαιωμάτων. Οι αλληλείς και αλληλευτική δυνατότητα είναι αυτοί που πρέπει να κερδίσουν. Και πιστεύω και συμφωνώ με τη συνάδελφο την κυρία Λεβίν ότι θα πρέπει να έχουμε ένα πιο μακρόπνο σχέδιο. Αλλά χωρίς αυτή την απειλή δεν υπάρχει μακρόπνο σχέδιο κατά με μπορούμε να ασχοληθούμε με τα θέματα διαχείρισης, με το ε, ΤΑΔΕ, με το ΔΙΝΑ, αλλά αυτή στιγμή δεν υπάρχει αυτή η απειλή της ίσης πρόσβασης σε ύδατα και πόρους που να σημαίνει ότι κάποιος άλλος μπορεί κάποιος να υποφοληθεί στο μέλλον από αυτά, δεν θα έχουμε καμία ελπίδα. Και ελπίζω να μπορέσουμε να το εξετάσουμε αυτό πριν καν αρχίσουμε να ασχοληθούμε τι με το τι μπορούμε να έχουμε αντί για ποσοστώσεις, ε, αν είναι ε, δυνατόν να εμπορευόμαστε δικαιώματα και ποσοστά και αν είναι καλή ιδέα. Εάν θέλετε να έχετε διαχείριση ελίας που θα είναι επιτυχημένη και νομίζω ότι όλοι αυτό θέλουμε, δεν μπορούμε να το καταφέρουμε εάν δεν δεχτούμε τη δήλωση ότι θα πρέπει να υπάρχει ίση πρόσβαση σε ύδατα και πόρους. Ο κύριος Μιλάνα. Για να σταθώ σε αυτά που μας είπατε να σταθούμε. Πιο ευχάριστο θα ήταν να κάνουμε μια γενική συζήτηση, αλλά τέλος πάντων για να τηρήσω αυτά που μας είπατε, εγώ θεωρώ ότι αυτά τα πέντε σημεία, αυτά τα πέντε άρθρα, αποδεικνύουν το εξής. Ε, δεν είναι πρόβλημα κύριε Κάντεκ, ε, σταματήστε. Λοιπόν, μας αποδεικνύουν το εξή. για το οποίο ε, δεν μπορώ να σιωπήσω. Συζητούμε την υποτιθέμενη νέα πολιτική αλίας, ξεκινώντας από το δεδομένο ότι οι προηγούμενες πολιτικές ήταν αποτυχημένες. Δεν μπορούμε να ξεκινούμε από αυτό το δεδομένο το έγγραφο στα πρώτα πέντε άρθρα δεν έχει ούτε κάτι καινούριο για την πολιτική, ούτε προϋποθέτει ότι γίνεται μία αντιστροφή στην πολιτική μας για το θέμα και ούτε καν δημιουργεί ή σχεδιάζει ένα μηχανισμό ο οποίος θα έπρεπε να απαντά με ε, καλό τρόπο στον όλο κλάδο, δηλαδή στην επιβίωση των αλλιέων και στη συμβίωσή τους με τα ψάρια. Και αυτό είναι το θέμα μας. Και η ανάλυση αυτών των πρώτων πέντε σημείων στο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν περιλαμβάνει κανένα στοιχείο το οποίο κατ' εμέ ε, να μας οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι είμαστε στο σωστό δρόμο για την ε, μεταρρύθμιση της κοινή ελευτικής πολιτικής. Θα πρέπει λοιπόν να συζητήσουμε αρχές. Όταν λέμε ότι πρέπει να ξεκινήσει το στάδιο της συμμετοχής στο σύστημα, ε, και των ενδιαφερομένων. Δεν μπορούμε να καθορίσουμε τις βασικές αρχές όταν ξέρουμε <coughs> τι θα αλλάξουμε σε σχέση με το παρελθόν. Η συμμετοχή δεν έχει κανένα νόημα εάν δεν συνοδεύεται και από κάποια υπόθεση συμμετοχής. Και ακόμα και η γενική παραπομπή στην περιφερειακή διάσταση δεν ε, καθορίζει κάτι καινοφανές, ένα νέο στοιχείο σχέσεων και διαχείρισης της διαδικασίας. Η μέγιστη βιώσιμη απόδοση, το MSY. Αυτό εξαρτάται από παράγοντες ε, βάσει των οποίων οργανώνεται το σύστημα. Και αν δεν θέλουμε να αλλάξουμε εκ βάθρων τις βασικές υποθέσεις στις οποίες εδράζεται το σύστημα, ουσιαστικά θα προσπαθούμε με γραφειοκρατικό τρόπο να τελειοποιήσουμε ένα μοντέλο το οποίο αποδείχθηκε στα τελευταία 20 χρόνια ότι είναι αποτυχημένο και μόνον. Θα μπούμε σε ένα φαύλο κύκλο. Θα αρχίσουμε σιγά σιγά να προσπαθούμε να τροποποιήσουμε εκείνο το άρθρο, εκείνο το άλλο άρθρο, αυτή την τάδε τροπολογία και δεν θα αλλάξουμε όμως τις τύχες και τις ε, προϋποθέσεις επιβίωσης του τομέα. Ήρεμα λοιπόν, λαμβάνοντα υπόψη ότι δεν έχουμε και πολύ χρόνο στη διάθεσή μα σήμερα, θα ήθελα να προτείνω το εξή στην κυρία Ρόντου, η οποία εργάζεται πολύ καλά προς αυτή την κατεύθυνση. Η πρότασή μου λοιπόν είναι η εξή. Όλο το οικοδόμημα στηρίζεται στο γεγονός ότι εμείς βλέπουμε το ψαρά και το ψάρι. Μετά βλέπουμε τα εργαλεία αλίας και τις ποσοστώσεις. Όλα αυτά βασίζονται σε αυτά τα τέσσερα θεμέλια. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε για τη θάλασσα ως αναπόσπαστο σημείο το οποίο έχει αφαιρεθεί από αυτή τη μεταρρύθμιση. Πουθενά δεν αναφέρεται η θάλασσα και ο σχεδιασμός του συστήματος. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο. Μπορούμε από εκεί και πέρα να ε, σκεφτούμε με όποια λογική θέλουμε. Αλλά αν δεν ξεφύγουμε από αυτή την παλιά λογική που έχει αυτές τις τέσσερις βασικές θεμελιώδεις αρχές, θα αρχίσουμε ε, μια ένα διαδικασία για να κάνουμε την ίδια δουλειά. Τον τρόπο με τον οποίο καθορίζονται οι ποσοστέωσει, το τάδε εργαλείο και όχι το άλλο εργαλείο, το τάδε πειραματικό στοιχείο, περιφερειοποίηση, ποσόστοση, πόση, τόση, λιγότερη, περισσότερη. Πρέπει πραγματικά να σκεφτούμε, στη χώρα μου λέμε βάζοντα ε, βάζοντας τα πράγματα στην άκρη. Προσπαθούμε να καταλογίσουμε τις άλλες προϋποθέσεις. Θα σας κάνω ένα ηλίθιο παράδειγμα που αφορά τη Μεσόγειο. Εμείς χρησιμοποιούμε ένα ε, σημαντικό μερίδιο των ε, ευρωπαϊκών ε, αποθεμάτων, κονδυλίων για το λεγόμενο αλλιευτικό απόθεμα. Δηλαδή, έχουμε δύο μήνες το χρόνο στους οποίους χρησιμοποιούμε πόρους, πληρώνουμε τους ψαράδες για να μην ψαράδι. κανείς. Πού? Πουθενά. Κλείνει η αλληλευτική περίοδος, οι αλληλείς κάθονται σπίτι τους, έχουν επιδοτήσεις για να μπορέσουν να επιβιώσουν και το λύσαμε το ζήτημα. Θεωρούμε ότι έχουμε δώσει μια απάντηση στην ε, κοινωνική ένταση που προκαλείται από, το, από την απώλεια εισοδήματο των αλλιών και θεωρούμε μέσα σε αυτούς τους δύο μήνες δημιουργούνται νέες βιολογικές συνθήκες και η θάλασσα είναι αυτή ε, η μηχανή παραγωγής αλλιευμάτων. Δεν ισχύει. Γιατί η πρώτη απάντηση καταρχά είναι ημοσύνη προς τους αλληλεί και η δεύτερη απάντηση είναι κοροϊδία, διότι για ένα ή δύο μήνες διακοπής της αλληλεία δεν αλλάζει τίποτα από βιολογικής πλευρά. Θεωρώ λοιπόν ότι θα έπρεπε αυτοί οι δύο μήνες διακοπής της αλληλείας σε όλους τους τομείς να μην είναι ένα κλείσιμο για τρία ή πέντε χρόνια του 20% της θαλάσσιας υποφέρειας στην οποία θα απαγορεύεται να δουλέψουμε. Για κανέναν. Δεν θα είναι γενική απαγόρευση, συνολική και να υπάρχει και ένα διάστημα στο οποίο θα δίνονται κίνοντρα στις χώρες ώστε να χρησιμοποιείται η θάλασσα ως απόθεμα και να θεωρήσουμε ότι είναι η μεγαλύτερη επιχείρηση ε, τροφοδότησης της θάλασσας. Έτσι είναι τα πράγματα. Αυτό είναι σαφέ. Αν κάθουμε να συζητάω τα τρία ή τέσσερα σημεία που μα παρουσιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η βαλίτσα πάει πολύ μακριά και δεν θα καταλήξουμε πουθενά. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να σταθούμε λίγο και να σκεφτούμε. Καταρχάς, να σκεφτούμε καταρχάς ω Ευρωπα... Επιτροπή και να κάνουμε και μια ειδική επιτροπή, κυρία Πρόεδρε, για το σκεπτικό μας, τη φιλοσοφία μας, το οποίο θα πρέπει να είναι συνέπεια αυτό που είπαμε στην Πράσινη Βίβλο. Υπάρχει και αυτό το σχιζοφρενικό σχεδόν σύστημα με το οποίο καταλήγουμε στη λήψη απόφασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση που νομίζω ότι θα πρέπει να σταματήσει, να σπάσει αυτός ο κύκλος. Κάναμε μια πράσινη βίβλο πριν από 1,5 χρόνο. Περιμένουμε διακαώ να ετοιμάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα έγγραφά τη και να περιμένουμε και μια πρόταση κανονισμού εμεί εδώ στο Κοινοβούλιο. Και εμεί που είμαστε Κοινοβούλιο και που στην μετά Λισαβόνα εποχή είμαστε αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να καθορίσουμε την πολιτική και να χαράσουμε την πολιτική εξακολουθούμε να κάνουμε τα μαθηματάκια μας στο τετράδιο και γράφουμε αυτά τα τέσσερα καθήκοντα, τα τέσσερις κανόνες που μας καθορίζει η ευρωπαϊκή πολιτική. Υπάρχουν δύο τρόποι να γίνει μεταρρύθμιση. Ή έχουμε ένα φουστάνι που έχει κάποια σκισμένα κομμάτια και θα βάλουμε μπαλώματα και για άλλα δέκα χρόνια θα έχουμε ένα μπαλωμένο φουστάνι ή θα αποφασίσουμε να γδυθούμε και να αντιθούμε με ένα καινούριο φόρεμα. Señor Σα Σας ευχαριστώ. Πρόεδρε. Δεν ξέρω κατά πόσο θα πρέπει να μιλήσω για συγκεκριμένους στόχους ή για τους γενικούς στόχους. Ο κύριος Μιλάνα ξεκίνησε μία πολύ συγκεκριμένη φιλοσοφική συζήτηση. Δεν ξέρω αυτός είναι ο στόχος μας. θα προστιμούσα να συγκεντρώσω την προσοχή μου σε ένα θέμα που θέλαμε να συζητήσουμε σήμερα, δηλαδή να εκφράσω την υποστήριξή μου για την ιδέα αυτή και να περιοριστούμε σε αυτά τα περιορισμένα τμήματα. Αυτό θα μας οδηγήσει ίσως σε φιλοσοφικές σκέψεις, αλλά θα μας επιτρέψει να ολοκληρώσουμε και την ε, συζήτηση. Η κυρία Ροντούσα αναφέρθηκε στι διαφορέ μεταξύ παραδοσιακή και βιομηχανική αλληλεία. Πραγματικά υπάρχει. Αναλύοντα το κείμενο του άρθρου 5 με τους ορισμούς, δεν υπάρχει ορισμός της ε, παράκτης αλίας και νομίζω θα πρέπει να σκεφτούμε κάτι τέτοιο σε ένα νέο ορισμό να σκεφτούμε μόνοι μας ή να στραφούμε προς επιστήμονες που θα μπορούσαν να μας δώσουν έναν ορισμό αυτού του τύπου της ελίας που μας ενδιαφέρει τόσο πολύ. Επίσης αναφερθήκαμε στην ε, περιφερειοποίηση. Στο άρθρο 4 σημείο 1 βλέπουμε την κατανομή μεταξύ των διαφορετικών επίπεδων ε, αρμοδιοτήτων, τοπικό, περιφερειακό, κρατικό, ευρωπαϊκό κλπ. Από τοπικής πλευράς υπάρχει πραγματικά μια διαφορά ή επειδή δεν ξέρουμε ακριβώ τι σημαίνει περιφερειοποίηση και προσπαθούμε να εφεύρουμε νέους όρους κινούμεθα προς την κατεύθυνση αυτή θα μπορούσαμε να σκεφτούμε και μακροοικονομικά ή μικροοικονομικά ή οτιδήποτε άλλο. Θα πρέπει νομίζω καλύτερα να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας στην ευρωπαϊκή πολιτική που είναι τμήμα των δικών μας αρμοδιοτήτων. Και στην περιφερειακή πολιτική θα πρέπει να προσθεθεί αυτό. Ευχαριστώ κύριο Γκάλαχερ. Πρόεδρε, εγώ δεν θέλω να γενικολογήσω, θέλω να αναφερθώ συγκεκριμένα στο σημείο της σημερινής διάταξης, πρώτο τμήμα. Ξέρουμε τις ε, απόψεις μας για την περιφερειοποίηση και θα πρέπει να βρούμε ποια είναι η λύση που μπορεί να βρεθεί σχετικά. Αρχίζοντας με το σημείο 5, και αυτά που αναφέρονται για την ε, βιώσιμη ανάπτυξη έχω να πω ότι ήμουνα το 2002 στο Ιωάννησπουργκ και αυτά που ακούγονται τώρα δεν είναι καινούργια, είναι ήδη στη δήλωση αυτή και στις ε, δυνατότητες εφαρμογής για το μέγιστο της ε, απόδοσης που θα πρέπει να είναι ο ακρογωνίος λίθος της ε, ε, αναθεώρησης. Και θα πρέπει να καλύπτονται οι στόχοι. Θα πρέπει όλα αυτά να εξεταστούν στις ετουλικές σκέψεις. Έχουμε εδώ μία απαγόρευση ε, να απαγορευτούν οποιοδήποτε ε, απορριψεις ε, αυτό δεν έχει νόημα. Θα πρέπει να δούμε κάποια κίνητρα καλύτερα. Και στο 23 που αναφέρεται η συνθήκη της Χάγης, υπό συγκεκριμένε προϋποθέσεις, όπως αυτές που τηρεί η χώρα μου κάθε χρόνο. Αυτό θα πρέπει να αναπτυχθεί καλύτερα στη διαφορά του. Δυστυχώ, για λόγους που γνωρίζει η Κομισιόν από μόνη τη, αποφάσισαν να μην μα δώσουν αυτό που είχαμε ζητήσει. Τώρα το 29 καλύπτει ε, τη δυνατότητα μεταφοράς των δεκτικών ε, ευκαιριών. Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό για ορισμένε χώρε. Ιδίω ο υποχρεωτικό χαρακτήρας είναι προβληματικό. Το Κοινοβούλιο και οι Επιτροπές μας συμφωνούν καταρχή ότι θα πρέπει κάθε κράτος μέλο να μπορεί να αποφασίσει ε, κατά πόσο κάτι τέτοιο θα είναι υποχρεωτικό ή όχι δεν προβλέπεται τίποτα όσον αφορά τις βιολογικά ευαίσθητες περιοχές, ως με η Ιρλανδική θάλασσα. Υπάρχει όμως η διάταξη 15 για τις Αζόρες, για τη Μαντέρα και για τις καναλίες νήσους. Γιατί η Ιρλανδική θάλασσα αποκλείεται από τις ε, βιολογικά ευαίσθητες περιοχές. Και κάτι άλλο, το θέμα των συμφωνιών με τρεις χώρες, στο 39 οι συμφωνίε αυτές θα πρέπει να καλύπτουν την ε, Νορβηγία, τις Φαρόε και την Ισλανδία. Αυτό είναι μια ε, σημαντική ανησυχία και επίσης λέγεται ότι θα πληρώνει η βιομηχανία για τον έλεγχο και στο 52 όσον αφορά τις ενισχύσεις θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν θα πρέπει οι αλληλείς να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις αποτυχίες των κρατών μελών. Επίσης, το σημείο 1β αφορά του τους βιολογικούς πόρους ε, γλυκού υδατός. Τα άρθρα 2 και 3 που καλύπτουν τα MSY ε, είναι σημαντικά. Αυτή είναι όμως συγκεκριμένη στόχη, όχι γενική, και θα πρέπει να ενταχθούν σε ε, στους συγκεκριμένους στόχους του άρθρου 3. Πρέπει να αναφέρουμε ότι υπάρχουν κάποιες δυνατότητες επίτευξης MSY για όλα τα είδη που αλλιεύονται στις μικτές, ε, στη μεικτή αλία ταυτόχρονα. Αυτό που λείπει από την πρόταση είναι μια αναφορά στο όπου είναι κάτι τέτοιο δυνατό που υπήρχε στην δήλωση του Johannesburg. συγκεκριμένη στόχη στο άρθρο 3 θα πρέπει να προβλέπεται η δυνατότητα αξιολόγηση των στοιχείων και θα πρέπει να, περι... να συμπεριληφθούν τα περιφερειακά γνωματικά συμβούλια ΡΑΚΑ στο 4 επίσης όσον αφορά το MSY και η προληπτική προσέγγιση στην διαχείριση της αλληλείας και των οικοσυστημάτων δεν είναι σωστές κατά τη γνώμη μου και θα πρέπει να επαναδιατυπωθεί. Να μην θεωρήσουμε λοιπόν ότι όλα ε, γράφηκαν ε, και είναι αδύνατο να τα αλλάξουμε. Χρειάζονται πολλές αλλαγές. Και σχετικά βέβαια με το σημείο 1, κατά την άποψή μου. Η κυρία Μπαραντίκα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να περιοριστώ σε αυτό που είπαμε και θα είμαι πολύ συγκεντρημένη γιατί ακούσαμε πάρα πολλά πράγματα ήδη. Να ξεκινήσω με το άρθρο 3, τους συγκεκριμένους στόχους. εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε καταρχά να κάνουμε μια αλλαγή και να αλλάξουμε το α με το γ, γιατί ο πιο βασικό στόχο κατά την άποψή μου θα πρέπει να είναι με τη μεταρρύθμιση αυτή να δημιουργήσουμε τι κατάλληλε συνθήκε, ώστε οι αποτελεσματικέ αλληλευτικέ δραστηριότητε, να είναι βιώσιμε και ανταγωνιστικέ. Από εκεί και πέρα μπορούν να έρθουν όλα τα υπόλοιπα, όπω η μείωση των ε, ανεπιθύμητων απορρίψεων, αλλά ο βασικό στόχο τη μεταρρύθμιση, κατά την άποψή μου θα πρέπει να είναι αυτό. και θα πρέπει να καθορίσουμε συγκεκριμένε συγκεκριμένες Δεύτερον, μιλώντας για την αρχή της οικονομικής διακυβέρνησης. Συμμερίζομαι τις ε, αρχές της χρηστής διακυβέρνησης ε, στη μεταρρύθμιση αυτή, και πιστεύω ότι θα πρέπει να δούμε λίγο την παράγραφο Β όταν μιλόμαστε για κατάλληλα μέτρα τα οποία θα βασίζονται στις καλύτερες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις. Τι σημαίνει οι καλύτερες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, δηλαδή ότι αποφασίζουμε θα πρέπει να γίνεται βάση επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, ναι, εντάξει, αλλά ποιες θα είναι οι καλύτερες, πώς γίνεται αυτό, χρειάζεται διευκρίνηση. Τρίτον, Αναφερόμαστε στην ανάγκη να υπάρχει και μια μακροπρόθεσμη προοπτική για τη χρηστή διακυβέρνηση. Ωραία, συμφωνώ, αλλά βάσει αυτού θα πρέπει να υπάρχουν και νέα άρθρα που θα βασίζονται και στα πολιετή σχέδια να αναφέρονται σε αυτά. Δεν αρκεί να έχουμε έναν ορισμό μόνο του τι είναι πολιετέ σχέδιο. Κατόπιν, ε, όπως σας είπα, θα πρέπει να υπάρχουν και άρθρα τα οποία θα πρέπει να καθορίζουν από τι θα αποτελείται ένα πολιετές ε, σχέδιο συνεχίζω με τη χρηστή διακυβέρνηση. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει ανάγκη για χρηστή διακυβέρνηση, η οποία θα πρέπει να ξεκινάει από κάτω προς τα πάνω και να μπορούμε να δημιουργήσουμε μια καλή μεταρρύθμιση και καλή διαχείριση των αρχών αυτής της μεταρρύθμισης από τοπικό επίπεδο, στη συνέχεια σε περιφερειακό και εθνικό για να φτάσουμε τελικώς στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Διότι για να αναλάβει τις ευθύνες του όλος ο τομέας και αν τις αναλάβει θα μπορέσουμε ίσως να βελτιώσουμε την κατάσταση μέσα αυτής της μεταρρύθμισης. Να πω επίσης ότι είναι απαραίτητο να αναφερθούμε και στην ερασιτεχνική αλληλεία. Θα πρέπει να υπάρχει ένας ορισμός του τι είναι ερασιτεχνική αλληλεία, διότι οι δυσκολίες και οι ανάγκες που έχουν οι παραδοσιακοί αλληλείς είναι διαφορετικές από τον πιο βιομηχανοποιημένο κλάδο. Επομένως θα πρέπει να υπάρχει ένας σαφής ορισμός του συγκεκριμένου αλληλευτικού κλάδου. Προσπαθούμε όλοι να βελτιώσουμε την κατάσταση. Θέλουμε να έχουμε ένα αλληλευτικό τομέα ο οποίος θα είναι βιώσιμος και ανταγωνιστικός ε, με κατάλληλη προστασία του περιβάλλοντος και του οικοσυστήματος όπως αναφέρουμε εδώ αλλά ταυτόχρονα θέλουμε η καλή κατάσταση της αλίας να μην συνδέεται άμεσα πάντα με τη ε, εισόδημα, διότι ε, υπάρχουν κάποια είδη τα οποία σταμάτησαν όταν βρίσκονται σε καλές συνθήκες και εκεί έρχεται η στιγμή όπου κάποιος θα αρχίσει να αποκομίζει κάποιο εισόδημα και ε, δεν υπάρχει καλή τιμή για το αλίευμα. Τα προβλήματα λοιπόν για τα εισοδήματα δεν ε, σχετίζονται μόνο με τις αλληλευτικές δυνατότητε, αλλά και σε άλλους τομείς. Αυτά λοιπόν ε, είναι σε γενικέ γραμμές αυτά τα οποία θα ήθελα να σχολιάσω. Η πρόεδρο. Θα κάνω και εγώ κάποιες μικρές παρατηρήσεις ξεκινώντα από το γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά. Θα περιοριστώ όμως τα πέντε άρθρα τα οποία υποτίθεται ότι συζητάμε σήμερα και θα ήθελα να κάνω τις εξής ερωτήσεις. Στο άρθρο 1, στο πεδίο εφαρμογή, θα ήθελε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μου εξηγήσει στο σημείο 1β εάν ε, η βοηλογική πόρη γλυκών υδάτων, διότι όπως είναι εδώ διατυπωμένο δημιουργεί κάποια σύγχυση, θα ήθελα να ξέρω αν τα θέματα της διαχείρισης και της εκμετάλλευσης ισχύουν για τους βιολογικούς πόρους γλυκών είναι λίγο συγκεχημένη η διατύπωση και δεν κατάλαβα αν εφαρμόζεται ή δεν εφαρμόζεται. Εγώ καταλαβαίνω ότι ισχύει, αλλά θα ήθελα να μου το διευκρινίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, στο άρθρο 1, στο πεδίο εφαρμογής, δεν αναφερόμαστε σε διαρθρωτική πολιτική και στις δυνατότητες του ελευτικού στόλου ή στις κοινέ οργανώσεις αγοράς, οι οποίες εμφανίζονται μόνο αργότερα σε κάποιο άλλο άρθρο και στις διεθνείς σχέσεις όταν στις αιτιολογικές εκθέσεις αναφέρεται ότι η εξωτερική πολιτική είναι αναπόσπαστο τμήμα της κοινή ελευτικής πολιτικής και δεν καταλαβαίνω γιατί δεν το περιλαμβάνετε όταν μετά στη συνέχεια στο διατακτικό το έχετε. Στο άρθρο 2 τώρα για τους γενικούς στόχους. Κατ' εμέ υπάρχει μία πρόβλημα στη διατύπωση μεταξύ του άρθρου 2, του γενικού στόχου και του άρθρου 3, των ειδικών στόχων. Νομίζω ότι στο άρθρο 2 θα πρέπει να έχει γίνει αναφορά στο άρθρο 30 ε, της συνθήκης. Πιο συγκεκριμένα το άρθρο 39, συγγνώμη, όχι 30, 39, γιατί υπάρχει η αρχή της ε, νομοθετικής ιεραρχίας. Καθορίζονται οι βασικοί στόχοι της κοινή αλληλευτικής πολιτικής και εκεί θεωρώ ότι με την περιορισμένη προοπτική που έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, επικεντρώθηκε μόνο στους περιβαλλοντικούς στόχους και λυσμόνισε και κοινωνικο-οικονομικούς ε, τομείς ε, που περιλαμβάνονται και αυτοί στο άρθρο 39. Δεν υπάρχει ισορροπία λοιπόν ούτε με το άρθρο 39 της συνθήκης ούτε ε, με τα άρθρα 9 και 8 της συνθήκης και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το έχουμε στους γενικούς στόχους ε, για τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση δεν θα πω τίποτα άλλο, τα είπαν οι συνάδελφοι και νομίζω ότι αυτό που αναφέρεται εδώ είναι η πιο ριζοσπαστική εναλλακτική λύση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την πιο ακρι... επέλεξε την πιο ακραία λύση σε αυτό το σημείο αυτό και νομίζω είναι αδύνατο να υλοποιηθεί ακριβώς και επειδή είναι ακραία και γι' αυτό το λόγο επιλέχθηκε. Στο σημείο 2, το είπε και η κυρία Λεβίνο, όταν λέμε ότι η εξμετάλλευση των ε, υδάτινων ε, πόρων μας επιτρέπουν να διατηρήσουμε τα επίπεδα άνω των επιπέδων που μπορεί να μας οδηγήσουν στη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Αυτό σημαίνει στην πραγματικότητα ότι ουσιαστικά θα ερμηνεύσουμε το MSY με πολύ περιορισμένο τρόπο και θα υποαλλιεύουμε, θα είμαστε κάτω από τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Επομένως νομίζω ότι δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο το έχουμε αυτό εδώ, διαφωνώ απολύτως με αυτό που αναφέρεται εδώ. Εγώ πιστεύω, όπως λέει και η αξιολόγηση αντικτύπου, ότι ορισμένα πιο ευέλικτα ε, στοιχεία τα οποία αναφέρονται θα πρέπει να αιτιολογούνται και να συγκεκριμενοποιούνται στα πολιετή σχέδια και δεν θα πρέπει να καθορίζονται στο άρθρο 2 και θα ήταν πολύ πιο λογικό για να μπορέσουμε να έχουμε και συνέπεια ε, με την ε, επιτυχία του ε, MSY. Πώς θα το εφαρμόσετε όμως ε, στην αλία πολλαπλών ειδών. Θα βασιστείτε ε, το ποσοστό του πιο, του πιο ακριβού είδους ή του αυτού που αλλιεύεται περισσότερο, πώς θα καθορίσετε τι γίνεται με, τα, ε, με την αλία πολλαπλών ειδών που είναι και κυρίαρχη μορφή αλίας στα ευρωπαϊκά είδατα. Στο σημείο 2 για τη Μεσόγειο, στο σημείο 15, αναφέρεστε σε ένα 20% μείωση της αλλιευτικής προσπάθειας ε, στη Μεσόγειο για τους γενικούς στόχους μας είπατε ότι, είπατε ε, ότι υπάρχουν και κάποιοι στόχοι που πρέπει να περάσουν στους γενικούς στόχους και να τροποποιήσετε το άρθρα 2 και άρθρα 3. Για το άρθρο 4 τώρα, αρχές της χρηστής διακυβέρνησης, στην πρώτη παράγραφο που αναφέρεστε στο σαφή ορισμό των ευθυνών σε ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, όπως είπανε πολλοί άλλοι, αυτό το άρθρο δεν έχει κανόνα νόημα γιατί το περιφερειακό στοιχείο δεν αναφέρεται πουθενά. Στην τρίτη παράγραφο, αν όντω χρειαζόμαστε ε, στις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις και τώρα το ποιες είναι οι καλύτερες επιστημονικές ε, γνωμοδοτήσεις δεν ξέρω ποιες είναι, ε, ποιες είναι οι καλύτερες και ποιος το αποφασίζει ότι είναι οι καλύτερες. Αλλά τέλος πάντων, ε, όσο περισσότερες και καλύτερες έχουμε, καλύτερε θα είναι τα αποτελέσματα. Αλλά το να θεωρούμε ότι είναι ουσιαστικά δόγμα, δεν νομίζω ότι ε, χρησιμεύουν σε τίποτα οι επιστημονικές νομοδοτήσεις αν τις αντιμετωπίζουμε ε, έτσι και δεν είναι αυτή η σωστή άγουσα. Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο είναι οι συνομοθέτες οι οποίοι αποφασίζουν βάσει των επιστημονικών νομοδοτήσεων για τη σωστή οδό. Στο σημείο σίγμα ΤΑΦ αναφερόμαστε στη συνοχή με την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική και τις άλλες πολιτικές της Ένωσης. Εγώ θεωρώ ότι η κοινή αλληλευτική πολιτική είναι τμήμα της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής. Δεν πρέπει να υπάρχει συνοχή. Είναι τμήμα της. Είναι λάθος η διατύπωση και επομένως ο προσανατολισμός που δίνεται δεν είναι ο κατάλληλος. Για το άρθρο 5... Δεν υπάρχει λόγος να αναφέρω τίποτα, είναι εκατοντάδες οι ορισμοί με τους οποίους διαφωνώ. Και θα ήθελα όμως να μου πείτε γιατί όταν καθορίζετε την οικοσυστημική προσέγγιση από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί επιλέξατε το συγκεκριμένο ορισμό όταν υπάρχουν και άλλοι ορισμοί που είναι δεσμευτικοί για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως για παράδειγμα τη Σύμβαση για την Βιολογική Ποικολομορφία ή υπάρχει και η Σύμβαση του 2002. Γιατί επιλέξατε αυτήν, ε, αυτόν τον ορισμό και όχι άλλε που κατά την άποψή μου είναι καταλληλότερε. Δεν θα σταθώ περαιτέρω στο θέμα αυτό, να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη συνέχεια συνέχεια στην κυρία Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Και σας ευχαριστώ για τα άφθονα και ενδιαφέροντα σχόλιά σας στην πρότασή μας. Δύο τεινά, λόγω του χρόνου που μου δίνετε στη διάθεσή σας. Ή θα τα σχολιάσω όλα και τα βασικά, ή αν δεν έχω αρκετό χρόνο, θα προσπαθήσω να απαντήσω όχι σε σχόλια ή σε απόψεις, αλλά μόνο στις ερωτήσεις που απευθύνθηκαν συγκεκριμένα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ, ε, κυρία Πρόεδρε, θα προσπαθούσα να απαντήσω ε, και να μην σχολιάσω παρατηρήσεις ή σχόλια, να απαντήσω στις συγκεκριμένε ερωτήσεις και αφού ολοκληρώσω, αν μου δώσετε και άλλο χρόνο, με τα χαράς να σας απαντήσω και στα υπόλοιπα. Καταρχάς, υπήρξαν αρκετές ερωτήσεις κυρίως από πλευρά της κυρίας Λεβίν, όταν αναφερόμαστε σε μέγιστη βιώσιμη απόδοση, αναφερόμαστε σε ε, βιώσιμη απόδοση από πλευράς βιομάζας ή από πλευράς θνησιμότητας. Και είναι σημαντικό αυτό. Αυτό όχι σε επίπεδο στόχου, αλλά σε επίπεδο ορισμού της εφαρμογής της αρχής της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης, η οποία θα εφαρμοστεί στην πολιτική διατήρηση των αποθεμάτων και στα μακροπρόθεσμα προγράμματα διαχείρισης. Η άγουσα που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα τελευταία χρόνια είναι πολύ συγκεκριμένη. Λέμε ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε στα μακροπρόθεσμα προγράμματα σε όρους θνησιμότητας αναείδος αλίας και όχι βιομάζας. Και γιατί αυτό. Απλώς και μόνον διότι η αυθονία της βιομάζας, ιδίως ε, η βιομάζα της μέχρι της βιώσιμης απόδοσης, προκύπτει από δύο παράγοντες. Από τη διατήρηση της αλίας, ε, τη διαχείριση συγγνώμη, της αλλά και από την ε, φυσικούς παράγοντες. Και επομένως μπορεί να καθορίσουμε εμεί ε, βιομάζα μέγιστης βιώσιμη απόδοσης, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιτύχουμε αυτό το στόχο. Εάν η φύση όμως δεν είναι ευνοϊκή στα συγκεκριμένα χρόνια, ό,τι προσπάθεια και να κάνουμε, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα καταφέρουμε να επιτύχουμε το στόχο αυτό. Το βασικό πλεονέκτημα της ε, θνησιμότητας ανά είδος αλίας είναι ότι αυτό είναι το στοιχείο που μπορούμε να ελέγξουμε και μπορούμε να διαχειριστούμε. Επομένως, αυτό που μπορούμε να κάνουμε στη διαχείριση της αλίας είναι να προσπαθήσουμε να διαχειριστούμε την θνησιμότητα αναλευτικό είδος, ώστε να προσπαθήσουμε να έχουμε τα λευτικά αποθέματα σε ένα συγκεκριμένο ποσοστό εκμετάλλευσης, τέτοιο το οποίο να μας επιτρέπει ώστε όποιο και να είναι το επίπεδο γενεοδορίας της φύσης, να πάρουμε το μέγιστο που μπορούμε να αποκομίσουμε από τη φύση για το συγκεκριμένο είδος εκμετάλλευσης. Επομένως, θέλουμε να επικεντρωθούμε σε αυτό που μπορούμε να διαχειριστούμε. Και η βιομάζα ε, νομίζω ότι είναι το καλύτερο παράδειγμα των αρχικών σχεδίων που είχαμε για τη Βόρεια Θάλασσα και το Βακαλάο εκεί. Καθορίσαμε κάποιους στόχους βιομάζας και μετά ε, ακόμα και η ίδια επιστημονική κοινότητα αντιλήφθηκε ότι ακόμα και αν σταματούσαμε να λιεύουμε, αυτοί οι στόχοι της βιομάδας θα ήταν αδύνατον να επιτευχθούν. Επομένως θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε πιο ε, ρεαλιστικούς στόχους για τους οποίους μπορούμε να έχουμε και κάποια επιρροή. Δεν μπορούμε να επηρεάσουμε τα ε, επίπεδα αυθονίας, αυτό το καθορίζει η φύση, αλλά μπορούμε να καθορίσουμε ποια είναι τα επίπεδα θνησιμότητας είδους, αναλευτικό είδους και αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Κατόπιν, υπάρχει μια ερώτηση, ως ερώτηση την εκλαμβάνω, γιατί πρέπει να υπάρχει αποκλειστική αρμοδιότητα, το είπε ο κύριος Χάτσον. Ε, κοιτάξτε, αν δεν το εξήγησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορώ να σας τα πω εγώ. Δεν θα επιμείνω πολύ σε αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ενδιαφέρεται να προτείνει καμία αλλαγή στο άρθρο 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου ε, καθορίζεται η αρχή ότι η διαχείριση των αλληλευτικών αποθεμάτων είναι αποκλειστική αρμοδιότητα. Σας διαβεβαιώ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει καμία πρόθεση να τα αλλάξει. Γιατί πρέπει να είναι αποκλειστική αρμοδιότητα. Γιατί τα αποθέματα είναι κοινά, τα αποθέματα που βρίσκουμε στα ύδατα οποιασδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κοινά αποθέματα τα οποία τα μοιράζεται με άλλε χώρε και εάν δεν είναι κοινά αποθέματα, εάν δεν γίνεται διαχείριση μέσω κοινή αλληλευτική πολιτική, τότε θα πρέπει να υπάρξει διαχείριση μέσω περιφερειακών οργανώσεων αλληλεία, τύπου τη ΝΕΑΦΚ, τη ΝΑΦΟ, τη ΆΙΚΑΤ. Και επομένω, σα ρωτώ, το μοντέλο διαχείριση αυτών των περιφερειακών οργανώσεων είναι πιο αποτελεσματικό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αφήνω το ερώτημα σε κρεμότητα. Μας ρώτησε επίσης ο κύριος Γκάλαχερ γιατί ε, στην πρόταση δεν αναφερόμαστε στην ε, βιολογικά ευαίσθητη περιοχή γύρω από την Ιρλανδία και αναφερόμαστε όμως στο καθεστώς περιορισμένης πρόσβασης ε, στις υπερπόντιες περιοχές των Καναρίων Νήσων, των Αζωρών και άλλων. Η απάντησή μου είναι η εξής η Μαδέιρα, οι Αζόρες και τα Κανάρια νησιά είναι θέματα καθεστώτος πρόσβασης. Ε, είναι θέματα τα οποία άπτονται του ελάχιστου καθεστώτος πρόσβασης των 100 μιλίων και των 12 μιλίων χωρικών υδάτων. Αυτές οι τρεις περιοχές, τα Κανάρια νησιά, οι Αζόρες και η Μαδέιρα, είναι υπερπόντιες περιοχές οι οποίες βάσει του άρθρου 349 της συνθήκης μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο πολιτικής θετικής διάκρασης ε, επειδή ακριβώς είναι υπερπόντιες περιοχές. Επομένως, το καθεστώς που ισχύει για τις Ασόρες, τη Μαδέιρα και τα Κανάρια νησιά δεν είναι τεχνικό μέτρο, είναι θέμα πρόσβασης, στο οποίο προτείνουμε συγκεκριμένη παρέκκληση στην αρχή της ελεύθερης πρόσβασης ε, στα 12 ε, ναυτικά μίλια ε, λόγω των συγκεκριμένων ε, χαρακτηριστικών των συγκεκριμένων αυτών περιοχών και δεν βασιζόμαστε σε καμία βάση στην κοινή πολιτική. Είναι μία βάση στην πολιτική θετικής διάκρισης για τις υπερπόντιες περιοχές οι οποίες καθορίζονται στο άρθρο 341 της συνθήκης. Να σας πω επίσης ότι η βιολογική ευαίσθητη περιοχή γύρω από την Ιρλανδία και ενό τελείω διαφορετικού καθεστώτος. Δεν πρόκειται για ένα μέτρο το οποίο αφορά την αρχή πρόσβασης, πρόκειται για ένα τεχνικό μέτρο προστασίας μιας ευαίσθητης περιοχής και η περιοχή ε, η οποία... Ε, συζητούμε είναι η Ιρλανδία, η οποία σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται υπερπόντια περιοχή. Είναι κάτι τελείω διαφορετικό. Γι' αυτό ακριβώ επιλέγουμε το συγκεκριμένο μέτρο και όχι ε, το άλλο μέτρο. Δεν προτείνεται καν η βιολογικά ευαίσθητη περιοχή στην Ιρλανδία, ούτε καν υπάρχει παρέκκληση. Υπάρχει ενισχύ η βιολογικά ευαίσθητη περιοχή, διότι δεν υπάρχει κάτι στην πρόταση που να δημιουργεί παρέκκληση ή να διατηρεί κάτι άλλο. Επίσης, ε, ε, αναφερθήκαμε στους ε, βιολογικούς πόρους γλυκών νερών και γιατί τους περιλαμβάνουμε εδώ. Το ίδιο ρώτησε και η κυρία Φράγκα και ο κύριος Γκάλαγκερ. Υπάρχει ένα πρόβλημα που έχουμε στον βασικό κανονισμό, το οποίο είναι ενισχύει αυτή τη στιγμή. Ο κανονισμός λέει ότι η κοινή αλευτική πολιτική χρησιμοποιείται στα ανάδρομα είδη στο Σολομό και στα κατάδρομα είδη στα, στα χέλια ε, στην περίοδο στην οποία ε, κυκλοφορούν σε γλυκά ύδατα. Γι' αυτό ακριβώς μπορούμε να έχουμε συγκεκριμένο καθεστώς και έχουμε ένα πρόγραμμα ε, ανασύστασης για τα χέλια. Όταν ε, συζητήσαμε το πρόγραμμα ανασύστασης για τα χέλια είχαμε πρόβλημα με τη νομική βάση. Πλέον διαθέτουμε νομική βάση που είναι ε, η κοινή ε, πολιτική και δεν είναι η βάση που έχουμε εδώ πέρα. Στη, για τα ανάδρομα και κατάδρομα είδη που έχουν ένα τμήμα του βιολογικού τους κύκλου σε γλυκά ύδατα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, να εφαρμόζουμε τη διαχείριση της κοινή ελευτικής πολιτικής. Αυτός δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε όλες τις διατέξεις της κοινή ελευτικής πολιτικής σε είδη τα οποία είναι αποκλειστικά γλυκών υδάτων. Υπάρχουν κάποια είδη γλυκών υδάτων στα οποία δεν ε, θέλουμε να έχουμε συγκεκριμένη διαχείριση ε, διότι αυτό αποκλείεται. Επαναλαμβάνω ότι η διάταξη έχει ως στόχο να καλύψει ανάδρομα και κατάδρομα είδη ε, και ε, είδη, τα είδη δηλαδή που έχουν τμήμα του βιολογικού τους κύκλου σε γλυκά ύδατα. Η κυρία Μπιλμπάου Μπαραντίκα ε, ρώτησε τι ακριβώς εννοούμε με τον όρο καλύτερες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις και γιατί το προτείνουμε. Αυτό που θέλουμε είναι η επιστημονική βάση ε, για την κοινιαλιευτική πολιτική γνωρίζουμε ότι δεν είναι τέλεια και δεν θα είναι ποτέ. Η επιστημονική βάση είναι πολύ σαφής. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις στις οποίες δεν έχουμε καν επιστημονικά στοιχεία και έχουμε και κάποιες φαιές ζώνες στις οποίες έχουμε μεν επιστημονικά στοιχεία αλλά δεν είναι τέλεια και είναι απλώς ενδεικτικά και λέμε απλώς ότι δεν μπορούμε όταν έχουμε ανεπαρκή επιστημονικά στοιχεία να το χρησιμοποιούμε ως πρόστιχημα για να μην ε, υιοθετήσουμε ε, μέτρα διαχείρισης όταν χρησιμοποιούμε και υιοθετούμε συγκεκριμένα μέτρα διαχείρισης, προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε το καλύτερο στοιχείο που έχουμε στη διάθεσή μας. Αυτό που προσπαθούμε λοιπόν είναι, επειδή οι επιστημονικές βάσεις μπορεί να είναι ατελείς, να μην χρησιμοποιείται αυτό ως πρόσχημα για να μην νομοθετούμε. Θέλουμε να έχουμε ένα υψηλό επίπεδο ε, προστασίας και επειδή δημιουργείται αβεβαιότητα πρέπει να τη διαχειριστούμε και πρέπει να τη διαχειριζόμαστε ακόμα και όταν δεν τα γνωρίζουμε όλα, όταν οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν τα πάντα, θα πρέπει να βασιζόμαστε σε αυτό το οποίο μας δίνουν οι επιστήμονες. Αυτό προσπαθούμε να πούμε με αυτή τη διάταξη. Κυρία Πρόεδρε, νομίζω ότι στην πρώτη ερώτησή σας απάντησα. Ε, με ρωτήσατε επίσης γιατί θέματα εξωτερικής ε, αλληλείας δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1. Το άρθρο 1 έχει ένα πεδίο εφαρμογής το οποίο ε, συμπεριλαμβάνει και αυτούς τους τομείς. Δεν τα αναφέρονται ρητά στη διατύπωση, αλλά εμείς θεωρούμε ότι καλύπτονται. Για το άρθρο 39, όπως είπατε και εσείς και νομίζω ότι πολύ καλά συνοψίσατε την κατάσταση, το άρθρο 39 της συνθήκης είναι πολύ ισορροπημένο. Ε, η πρόταση ε, λέτε ότι δεν είναι, σε αυτό διαφωνώ. Θα πρέπει να είμαστε πολύ σαφείς εδώ και νομίζω ότι όλες οι παρεμβάσεις που ακούσαμε με τον ένα με τον άλλο τρόπο αναφέρθηκαν σε αυτό το σημείο. Αυτό που προτείνουμε είναι απόλυτη ισορροπία μεταξύ περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών πτυχών. Το θέμα είναι πού βρισκόμαστε στο σημείο αυτό. Και νομίζω ότι αυτά είναι ουσιώδη. Είναι ίσως και το πιο ουσιώδη ζήτημα του πρώτου κεφαλαίου. Όπω είπατε και εσείς κυρία Πρόεδρε, το άρθρο 39 της συνθήκης καθορίζει μια σειρά από στόχου που δεν έχουν ε, κάποια ιεράρχηση συγκεκριμένη. Ορισμένες φορές είναι αμοιβαία αποκλειστική, ορισμένες φορές είναι συμβατά, ε, αλλά δεν υπάρχει συγκεκριμένη ιεραρχία. Το λένε όλοι και θα πρέπει να κάνουμε ε, ό,τι μπορούμε προκειμένου να επιτύχουμε όλους αυτούς τους στόχους από κοινού. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε και το έχουμε και στο βασικό κανονισμό, στον 2371 του 2002, οι συγκεκριμένοι στόχοι του άρθρου 39 της συνθήκης να συνδυαστούν με τους ε, στόχους αυτούς τους περιβόητους της βιώσιμότητας από κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής σκοπιάς. Ε, εμείς θέλουμε να έχουμε ισορροπία, αλλά το πρόβλημά μας είναι ότι μπορεί κάλλιστα να υπάρξει κάποια στιγμή όπου να υπάρχει απόλυτη ισορροπία και μεταξύ των τριών η μέγιστη βιώσιμη απόδοση κατ' εμάς είναι ό,τι πιο εγκύτερο έχουμε σε αυτή την ισορροπία. Το πρόβλημα είναι η μετάβαση στις περιπτώσεις στις οποίες είμαστε μακράν ε, της ισορροπίας. Τι κάνουμε για να την επιτύχουμε επειδή λέμε ότι θέλουμε να έχουμε ισορροπία μεταξύ αυτών των τριών ε, στόχων, στην πραγματικότητα, και σας το λέω γιατί εδώ και τρία χρόνια καθορίζω τα τάκια της ποσοστώσης, η ισορροπία μεταφράστηκε τελικώς στην πλειονότητα των περισσοτώσεων σε προτεραιότητα, σε κοινωνικο-οικονομικές ε, πτυχές βραχυπρόθεσμες. Και όλη η ιστορία της κοινή ελευτικής πολιτικής είναι ακριβώς αυτό. Οι κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες βραχυπρόθεσμα ήταν αυτές οι οποίες κυριάρχησαν όταν έπρεπε να λάβουμε υπόψη ε, τα στοιχεία που έπρεπε να λάβουμε και όχι η βιολογική και περιβαλλοντική στόχη μακροπρόθεσμα. Αυτό λοιπόν που ε, συμβαίνει και αυτό το οποίο ε, εξάγω εγώ συμπέρασμα είναι ότι δεν ήταν ισορροπημένη και ήταν πάντα υπέρ των κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων που είχαμε και μάλιστα των βραχυπρόθεσμων. Θέλουμε λοιπόν να έχουμε μία προϋπόθεση η, την επίτευξη των περιβαλλοντικών και βιολογικών στόχων ως προϋπόθεση για να μπορέσουμε να επιτύχουμε την ισορροπία. Αυτή είναι λοιπόν η, ισορροπία, η φιλοσοφία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μπορούμε να έχουμε ισορροπία μόνο εάν έχουμε ως προϋπόθεση την ανασύσταση των βιολογικών αποθεμάτων. Αυτό είναι ε, το οποίο υφέρπει της φιλοσοφίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το γεγονός ότι ο στόχος ε, μπορεί να είναι ανώτερος της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης και ότι αυτός ο στόχος είναι υπερβολικός. Κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να σας υπενθυμίσω εδώ ότι η μέγιστη βιώσιμη απόδοση και η αλληλεία δεν είναι ακριβείς επιστήμες, δεν είναι μαθηματικά. Για τους στόχους, όσο καλά και να τους καθορίσουμε από πλευράς θνησιμότητας αναλυευτικό είδους, είμαστε πάντα κατά προσέγγιση, είμαστε γύρω από το στόχο μας. Ε, η μέγιστη βιώσιμη απόδοση ε, έχει ως εξή. Η φύση ποτέ δεν θα μας καθορίσει τα πράγματα κατά τρόπον ώστε να πούμε ότι κοιτάξτε να δείτε να το σωστόχο μας τον επιτύχαμε. Εάν υπάρχουν διακυμάνσεις θα πρέπει να υπάρχει ένα κάποιο επίπεδο περιθώριο ασφαλείας το οποίο να μας επιτρέπει να πούμε ότι είμαστε σταθερά σε επίπεδο μέγιστης βιώσιμης απόδοσης και δεν έχουμε σκαμπανεβάσματα πάνω κάτω. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να προσπαθήσουμε αυτή η μέγιστη βιώσιμη απόδοση να μας επιτρέπει να έχουμε μια κάποια διακύμανση ώστε να είμαστε γύρω από το στόχο μας. Γι' αυτό λέμε ότι θέλουμε να, να είμαστε πάνω από τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Γιατί μέγιστη βιώσιμη απόδοση και την αλία πολλαπλών ειδών. Ε, κύριε Πρόεδρε, αύριο το πρωί έχουμε ειδική συνεδρία ακριβώς για αυτό το θέμα. Νομίζω ότι μπορούμε να το συζητήσουμε αύριο το πρωί ακόμα καλύτερα. Για το γεγονός ότι οι επιστημονικές γνωμοδοτήσεις είναι δόγμα και επιβάλλονται, διαφωνώ. Ε, το είπατε εσείς κυρία Πρόεδρε, δεν θα πρέπει να είναι δόγμα. Θα πρέπει να επενθυμίσουμε εδώ όμως ότι κάποια άλλα συστήματα, όπως για παράδειγμα το σύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών που αναφέρθηκε, ε, ο νόμος εκεί υποχρεώνει να ακολουθούνται επιστημονικές νομοδοτήσεις. Εδώ όμως δεν έχουμε ένα σύστημα ε, όπου είναι δόγμα αυτό που λένε οι επιστήμονες. Αν είχαμε το αμερικανικό σύστημα τότε ναι, αλλά εμείς δεν έχουμε αμερικανικό σύστημα. Κυρία Πρόεδρε, να ρωτήσω το εξή. Έχω άλλο χρόνο για να συνεχίσω να μιλάω ή να σταματήσω εδώ. Τι να σας πω. Εγώ θα προτιμούσα να συνεχίσετε εσείς, αλλά δυστυχώς πρέπει να κάνω συνεδρία συντονιστών. Δεν μπορώ να κάνω καλύτερη κατανομή του χρόνου από αυτό που έκανα. Από τούδε και στο εξή θα πρέπει να αφιερώνουμε περισσότερο χρόνο για τα θέματα αυτά. Δυστυχώ σήμερα πρέπει να σταματήσω γιατί έχουμε συνεδρία των συντονιστών Αύριο έχουμε ακρόαση και το πρωί και το απόγευμα. Πραγματικά πρέπει να γίνει συνεδρία των συντονιστών σήμερα. Δεν μπορώ να του βάλω αύριο. Αύριο το απόγευμα θα προσπαθήσουμε να συζητήσουμε τις εκκρεμότητες. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Ρόντας, θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο-τρία λόγια μόνο. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω όλους οι οποίοι συμμετείχαν στη συζήτηση και είδα ότι αυτό που είπα βασικά έγινε δεκτό από όλους. Θα ήθελα όμως να παρακαλέσω να τηρήσουμε τα θέματα που είχαμε συμφωνήσει, γιατί αλλιώς περιπλέκουμε περιτά και δεν θα μπορέσουμε να τηρήσουμε και το χρονοδιάγραμμα που είχαμε ορίσει. Θα ήθελα να μπορέσω να απαντήσω και συγκεκριμένε ερωτήσει. Τι ρώτησε για το χρονοδιάγραμμα. Εγώ θεωρώ ότι τον Ιούλιο θα πρέπει να υιοθετήσουμε την έκθεση αυτή στην Επιτροπή μα και να περάσουμε στην Ολομέλεια του Σεπτεμβρίου. Εάν όμω κάθε φορά συζητάμε όλα τα θέματα δεν θα τα καταφέρουμε. Και γι' αυτό ακριβώ είχαμε συμφωνήσει να εξετάσουμε σήμερα μόνο τους στόχους και το MSY. Εγώ δεν είπα τίποτα για την περιφερειακή τύχη, ούτε τα, όσον αφορά τα μέσα αλίας ε, και θα πρέπει να τηρούμε αυτό που είχαμε συμφωνήσει. Έχοντας ακούσει τους συναδέλφους νομίζω ότι θα μπορέσουν από κοινού να πετύχουμε μια λογική λύση ή μια πολιτική ισορροπημένη, γιατί νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Η παλαιότερη αλληλευτική πολιτική ήταν εν μέρη καταστροφική. Θα πρέπει να βελτιώσουμε και νομίζω ότι έχουμε μεγάλη ευθύνη και για τον τομέα και για τους απογονούς μας και για την οικολογία. Και θα πρέπει να φροντίσουμε όλοι αυτό να γίνει κατανοητό από τους ενδιαφερόμενους και τους συμμετέχοντες. Σας ευχαριστώ. Όλοι συνέβαλαν σημαντικά και στην επόμενη συζήτηση θα προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πριν ξεκινήσουμε τη συνδυασία των συντονιστών, να σα πω ότι χρειάστηκε να αλλάξουμε την ημερήσια διάταξη. Αύριο από 9 ω 9.30 θα συζητήσουμε την έκθεση Φεραίρα που είχαμε προβλέψει για σήμερα. 9.30 θα έρθει η υπηρεσία ελέγχου. Ε, μετά θα έχουμε τον κύριο Ρωμέβα Ιρουέδα για τον ερυθρό τόνο και μετά τα επόμενα σημεία μέχρι το 14 και το 15 και το 16 αν δεν υπάρχει χρόνος θα τα αναβάλουμε για άλλη μέρα γιατί ήταν ενημερωτικά από μένα. Ευχαριστώ. Άρε, ε, πέρασε η συνεδρίαση και θα ήθελα να ζητήσουμε ε, μόνο στους συντονιστές να παραμείνουν στην αίθουσα.